μας έχει ζητήσει κάτι ο κύριος Χάγκλον. Ε, Σαν 3α μικρό στην ημερήσια διάταξη. Νέα συμφωνία σύνδεσης με την Κινέα Μπισάου. Θα πρέπει λοιπόν να δεχθούμε το αίτημα αυτό μετά από την παρουσίαση της έκθεσής του για το Μαρόκο. Έχει ζητηθεί επίσης και από την κυρία Τρότμαν να παρουσιαστεί από την Επιτροπή για την οποία προετοιμάζει εν πάση περιπτώσει μια γνωμοδότηση σχετικά με την Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους θα υπάρξει αναβολή. Με αυτές τις τροποποιήσεις ελπίζω ότι γίνεται δεκτή η μερίσια διάταξη. Σαν πρόεδρο δεν έχω να ανακοινώσω τίποτα. Περνάμε λοιπόν στο 3 αμέσω. Συμφωνία με το Μαρόκο. Χακλούντ. Όλοι είχατε τη δυνατότητα να διαβάσετε την έκθεσή του. Του δίνω το λόγο. Κύριε Χάκλοντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Οι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε καλά. Λόγω ορισμένων δραστηριοτήτων συναδέλφων, το θέμα αυτό έχει ήδη αναβληθεί αρκετές φορές, αλλά έχει συζητηθεί και στην τελευταία Ολομέλεια, όπου υπήρξε ψηφοφορία και γι' αυτό ξαναρχόμαστε στη συζήτηση. Μιας και η πλειοψηφία δεν αποφάσισε, εν πάση περιπτώσει, να αναπέμψει το θέμα, το θέμα τίθεται στην ημερήσια διάταξή μας σε κανονική βάση και θα συνεχίσουμε ουσιαστικά τη συζήτηση την οποία είχαμε ξεκινήσει στο παρελθόν. Για πάρα πολλούς συναδέλφους το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερα πολιτικό. Εγώ σαν εισηγητής περιορίζω την προσοχή μου στη συγκεκριμένη συμφωνία, λαμβάνω υπόψη τις οικολογικές και οικονομικές διαστάσεις χωρίς να παραγνωρίζω βέβαια ότι η συζήτηση η οποία θα γίνει στα πλαίσια της μικτής κοινοβουλευτικής είναι μια συζήτηση η οποία έχει βαθιά πολιτικό χαρακτήρα. Κάτι το οποίο δεν κάνει τη δουλειά μου πάρα πολύ εύκολη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω για τους συναδέλφους να μπορέσουμε να το δούμε το θέμα σαν αλλιευτική συμφωνία πάντως κυρίαρχα. Η εταιρική σχέση με το Μαρόκο είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η μεγαλύτερη από τις χώρες εταίρους σε αυτή την κατηγορία που θέλουμε να υπογράψουμε ε, μια τέτοια συμφωνία. Και τώρα και στο μέλλον, ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουμε, το θέμα είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Επί της συμφωνίας αυτής. Um, I'm, Με πάρα πολύ λύπη και με πάρα πολύ ανησυχία διάβασα την έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης η οποία λέγει ότι η συμφωνία ήταν ε, απογοητευτική δεν επηρέασε τον τομέα της αλίας ε, στο Μαρόκο ούτε και σε επίπεδο ζήτησης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά είναι κάτι που λειτουργήσε εις βάρος του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Γενικά δεν είναι μια επιτυχής συμφωνία. Όλα αυτά τα έχω πει και στο παρελθόν όταν συζητούσαμε τα θέματα αυτά και δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω. Εγώ είχα αρκετές επικοδομητικές και θετικές συζητήσεις με τις αρχές του Μαρόκου με τον πρέσβη, ο οποίος ε, με αναζήτησε, συζητήσαμε μαζί και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φυσικά για το αν τώρα η έκθεση αξιολόγησης είναι σωστή ή όχι, να πω ότι στα πλαίσια των ανταλλαγών επιστολών με την πλευρά του Μαρόκου ε, ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα της ε, εκ των αξιολόγησης. Πολλοί πίστευαν ότι, έχουν διαβάσει μια, ότι είχαν διαβάσει μια διαφορετική εν πάση περιπτώσει ε, έκθεση. Οι Μαροκινοί φυσικά λέγουν ότι τα ευρήματα της ε, έκθεσης αυτής δεν είναι σωστά. Ασκούν κριτική στην έκθεση αυτή. Το υποστηρίζουν αυτό, αλλά εγώ περιμένω κάποια δεδομένα για να το αποδείξουν. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, δεν πήρα τέτοιου είδους δεδομένα. Αν κάποιος από εσά θέλει πράγματι να πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης, τότε είμαι στη διάθεσή σας να μου δώσετε στοιχεία και επιχειρήματα. Ακούγονται πολύ τις τελευταίες εβδομάδες τέτοιου επιχειρήματα διαδρομικά αλλά για να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα στη διάθεσή μας, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε. Λοιπόν, τα ευρήματα της έκθεσης εκ των υστέρων αξιολόγησης είναι ιδιαίτερως ανησυχητικά, Πρόεδρε. Και αυτό με οδηγεί στο να πω ότι αν πράγματι το Κοινοβούλιο παίρνει σοβαρά τον εαυτό του και τις υποχρεώσεις που έχει στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, αναλαμβάνουμε την αποστολή να εξετάζουμε τις εκθέσεις αυτές, να υπογραμμίζουμε τις δυσκολίες και αν πράγματι θέλουμε σοβαρά να αξιολογήσουμε την ισχύουσα συμφωνία στον τομέα της Αλίας με το Μαρόκο, είναι καθήκον μας να δράσουμε πλέον. Ταυτόχρονα γνωρίζω ότι πολλοί θα υποστηρίξουν ότι δεν μπορούμε να πούμε ναι ή όχι στην ερώτηση αν είναι καλή ή όχι η συμφωνία. Και μπορούμε ίσως να διορθώσουμε κάποια από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και στα πλαίσια των συμπληρωματικών πρωτοκόλων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ίσως, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί στα πλαίσια των επεξεργασιών για τη νέα συμφωνία μετά από το μήνα Φεβρουάριο. Να πούμε λοιπόν ότι εγώ δεν είναι ότι δεν θέλω να σταματήσουμε να έχουμε κάποιες αλλιευτικές συμφωνίες με το βασίλειο του Μαρόκου μόνο και μόνο επειδή σε ορισμένες πλευρές η παρούσα συμφωνία δεν είναι ικανοποιητική για μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία. Θα έχουμε και μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι μπορούμε να κάνουμε για να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη συμφωνία με το Μαρόκο. Και το Μαρόκο θέλει με επικρατηματικό τρόπο να προχωρήσουμε σε μια τέτοια συμφωνία. τέλο. κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι το θέμα αυτό είναι πολιτικά ιδιαίτερο ευαίσθητο αλλά όλο αυτό το δράμα γύρω από τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει να μην μας ε, τρομάξει. Να πω ότι ήδη από το 89, από το 99 συγγνώμη, πάνω από 12 χρόνια δεν είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία με το Μαρόκο. Για 8 χρόνια δεν υπήρξε μια συμφωνία και δεν υπήρξε και κανένα τρομερό πρόβλημα και από τις δύο πλευρές. Δεν θα πρέπει συνεπώς να να υπερβάλλουμε για τις πιθανές συνέπειες της περίπτωσης ε, κατά την οποία θεωρεί ότι η συμφωνία το κοινοβούλιο δεν είναι καλή και δεν τη δεχτεί. Παρ' όλα αυτά αυτό με ανησυχεί το τι θα γίνει με τους αλληλείς και με τις αλλιευτικές δραστηριότητες στο Μαρόκο και γύρω από τις ακτές του Μαρόκου. Θα χρειαστούν δύο μήνες για να περάσουμε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να τερματιστεί η συμφωνία αυτή. Έτσι και αλλιώς θα τερματιστεί γιατί έχουμε, ξεπερνάμε στο τέλος του μήνα την παράταση κατά ένα έτος και τα περισσότερα αλλιευτικά δικαιώματα για την περίοδο αυτή παράτασης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει αφού έχουν καταναλωθεί θα πρέπει να δούμε με την ψηφοφορία το Δεκέμβριο που θα καταλήξουμε. Αλλά τα περισσότερα πλοία ήδη μέχρι τότε θα έχουν αποσυρθεί γιατί έχουν εξαντλήσει τις ποσοστώσεις τους. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει λοιπόν ότι η κατάσταση είναι πράγματι δραματική στην περίπτωση κατά την οποία δεν συνενέσουμε. Να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι έχουμε μια μεγάλη ευθύνη εδώ να προστατεύσουμε τον φορολογούμενο, αλλά να είμαστε φιλικοί και για το περιβάλλον και ειλικρινείς απέναντι στους πολιτικούς μας εταίρους. Έχουμε σκεφτεί το θέμα αυτό πάρα πολύ, έχουμε ξενυχτήσει πάρα πολύ. Όσο το εξετάζουμε τόσο πείθομαι τελικά ότι μια τέτοια συμφωνία δεν είναι καλή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό ακριβώς σας προτείνω να μην συνενέσουμε στην εταιρική αυτή συμφωνία αλληλίας με το Μαρόκο. Και αυτό που είπα δεν είναι πολιτική δήλωση σε καμία περίπτωση πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω είναι εξαιρετική αυτή η συμφωνία, όχι μόνο γιατί καταλαμβάνει πάνω από ένα τέταρτο των κονδυλίων που έχουμε για όλες τις ε, συμπράξεις και δεν πετυχαίνει τίποτα. Ούτε για μας, ούτε και για τους Μαροκινούς. Οι Μαροκινοί έχουν ε, ένα μεγάλο αλλιευτικό στόλο, μεγαλύτερο από της Ισπανίας και της ε, Γαλλίας σε ό,τι αφορά το τονάζ και αλλιεύουν το 99% των δικών τους των και εξάγουν μεγάλες ποσότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι επιδοτούμε μερικούς αλληλείς σε μεγάλο βαθμό και αυτό που κάνει εξαιρετικά ε, ε, αυτή την έκθεση είναι η, ότι η αξιολόγηση καταλήγει λέγοντας ότι αναποτελεσματικότητα αυτής της συμφωνίας την ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Για το φορολογούμε της Ευρώπης αυτή είναι μια πολύ πολύ κακή συμφωνία και θα πρέπει να την τερματίσουμε. Ευχαριστώ κυρία Λόβιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βασικά συμφωνώ με αυτό που μόλις είπε τώρα ο κύριος Δέβης είναι μια συμφωνία που δεν συνεισφέρει και πολύ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και στο Μαρόκο. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι θα πρέπει να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει συμφωνίες αλίας μόνο με χώρες ε, οι οποίες έχουν πλεόνασμα αλλιευμάτων και η αξιολόγηση δείχνει ότι όλα τα αποθέματα είναι είτε ε, πλήρως, έχουν πλήρως ε, εκμεταλλευτεί εκτός από ένα απόθεμα που είναι στο νότο και που ανήκει στα, στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας. Αλλά η πρόσθετη εκμετάλλευση αυτού του αποθέματος θα σημαίνει υπερεκμετάλλευση λούκιου και άλλων ειδών. Ε, επίσης δεν υπάρχει κοινή διαχείριση αυτών των αποθεμάτων με άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής και υπάρχει υποψία ότι ίσως να υπάρχει υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων. Ε, το, η συνιστόσα ανάπτυξης αυτής της ε, συμφωνίας επίσης ε, δεν αποτελεί τίποτα και αυτό που οι ήδη Μαροκινοί δηλώνουν ότι τομεακή στήριξη που δίνεται στο Μαρόκο χρησιμοποιήθηκε μόνο κατά 15%. Αυτό είναι 0,2% των συνολικών επενδύσεων στον τομέα αλίας από το 2008 μέχρι το 2010. Και ο στόχος της πολιτικής του Μαρόκου είναι να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή του. Και έτσι πρέπει να γίνει. Και και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε καλοί γείτονε και να μην ασκούμε ε, πιέσεις ή να συνεχίζουμε συμφωνίες που να διακυβεύουν την ε, αηφορία του περιβάλλοντος και να μην ε, συνεισφέρουν την βιωσιμότητα του Μαρόκου. Αλλά επίσης, επειδή ο εισηγητής θέλει να τονίσει ότι δεν κάνει πολιτική δήλωση, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στην πολιτική κατάσταση που αποτελεί το υπόβαθρο αυτής της ε, προσωρινής συμφωνίας ε, που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και αν θυμάστε, είχαμε την νομική γνωμοδότηση από το την νομική υπηρεσία του ΔΕΚ που παρουσιάστηκε σε αυτή την Επιτροπή και στην Επιτροπή Ανάπτυξη το 2009. Εκείνη η γνωμοδότηση έλεγε ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επειδή η Δυτική Σαχάρα που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία ε, δεν είναι επικράτεια ε, που έχει την κυριαρχία της, εάν το Μαρόκο έχει το δικαίωμα να πολύ ε, ψάρια στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα ωφέλη ε, των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας. Από το 2009 η Επιτροπή, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, προσπάθησε να ε, εξασφαλίσει μια απάντηση από το Μαρόκο σε αυτό το ερώτημα. Πρώτη προθεσμία, αν θυμάμαι σωστά, ήταν ε, Αύγουστος του 10 από πλευρά της Κομισιόν να, ε, για να έχουμε κάποια χρονοδιαγράμματα να αξιολογηθεί η απάντηση του Μαρόκου. Το Μαρόκο όμω δεν έδωσε την απάντηση πριν από τις 13 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, που ήταν δύο μήνες πριν από την ε, διευρεύνηση αυτής της συμφωνίας. Δεν είχε η Κομισιόν αρκετό χρόνο να αξιολογήσει λοιπόν αυτή την απάντηση. Είδα την απάντηση. Είναι σε μορφή παρουσίασης PowerPoint. Μπορείτε να την ελέγξετε αν θέλετε ε, στην γραμματεία της Επιτροπής ΠΕΣ. Δεν γνωρίζω ακριβώς ε, τι θέλει να αξιολογήσει η Κομισιόν από αυτά τα γεγονότα, διότι είναι πολύ επιφανειακή. Είναι απλά μια περιγραφή της αλληλευτικής πολιτικής του Μαρόκου και δεν αναφέρεται καθόλου στη Δυτική Σαχάρα, μόνο ε, γεωγραφικές ενδείξει γίνονται. Άρα, το Μαρόκο έχει συμβάλει σε αυτή την περίπλοκη κατάσταση και θέλω να κλείσω λέγοντας ε, ότι συμφωνώ με τον εισηγητή ότι υπό αυτές τις περιστάσεις δεν πρέπει να δώσουμε τη συνένεσή μας αυτή την συμφωνία. Ευχαριστώ. Μπορώ να σας ζητήσω να είσαστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι, γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι. Ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια σε σχέση με αυτά που είπε και ο εισηγητής και οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις τουλάχιστον λόγια για να μην δώσουμε την έγκρισή μας τη συγκατάθεσή μας για αυτή τη συμφωνία. Ο ένας αναφέρθηκε σαφώς, ο οικονομικός, και είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση τώρα στην Ευρώπη οικονομικά και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να δεχτούμε κάτι που σε οικονομικούς όρους θα είναι απόλυτα ανεπαρκές. Δεύτερο λόγο οικονομικό, οικολογικό, συγγνώμη, και αυτό είναι σαφή. Συμφωνούμε με τι αξιολογήσει που έχουν γίνει για τα αποθέματα. Όντω είναι πολύ κακή ή κακή η κατάσταση των αποθεμάτων. Οπότε θα πρέπει αυτό να μα ανησυχήσει. Δεν μπορούμε απλώ να πούμε ότι α, δεν συμβαίνει αυτό, δεν ισχύει. Πρέπει να είναι σαφέ και να πούμε ότι μα ανησυχεί. Και ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το πούμε αυτό είναι μη δίνοντα τη συγκατάθεσή μα για την συμφωνία. Ο τρίτος ε, λόγος, επίσης ε, ακούστηκε από την ε, συνάδελφο, είναι ο πολιτικός λόγος. Για την πολιτική κατάσταση έχω να πω δύο πράγματα. Αυτή η συμφωνία μιλά για ένα κομμάτι της επικράτειας που δεν είναι κυρίαρχη, όπως ας πούμε τα είδατα στη Δυτική Σαχάρα. Πρέπει να πω καταρχάς ότι η Επιτροπή ζητά επανειλημμένως από τους Μαροκινούς να τους δώσουν πληροφορίες για το πώς πληρεί τι προποθέσει και τα συμφέροντα της δυτικής, του πληθυσμού τη Δυτική Σαχάρα αυτή η συμφωνία. Αυτέ οι πληροφορίε πάντα έρχονταν αργά και πάντα ήταν πολύ περιορισμένε. Αυτό που δεν έκανε μέχρι τώρα η Κομισιόν, από όσο ξέρω εγώ, είναι να ζητήσει να μάθει ποιε είναι οι επιθυμίε του πληθυσμού τη Δυτική Σαχάρα. Να μιλά δηλαδή για ε, νομιμοποιημένο εκπρόσωπο αυτή τη περιοχή. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει νομιμοποίηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ω. προς αυτό. Και επίσης ήδη υπάρχουν άλλες συμφωνίε με το Μαρόκο, με τι ΣΥΠΑ με τις χώρες ε, ε, που, ε, ε, ε, ελεύθερο εμπορίο που σημαίνει ότι μπορούμε να εντάξουμε τη συμφωνία αυτή σε αυτές τις συμφωνίες. Τουλάχιστον μπορούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αποκλείσει τη Δυτική Σαχάρα και τα ε, ύδατά της από τη συμφωνία αυτή, που επίσης μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, από όσο ξέρω τουλάχιστον, έχει προταθεί, αλλά δεν έχει εγκριθεί από την Κομισιόν. Οπότε αυτό πολιτικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δεχτούμε. Η συζήτηση που κάναμε πρόσφατα για το κατά πόσο θα πρέπει το θέμα αυτό να πάει στο δικαστήριο δείχνει ότι αυτό το θέμα εξακολουθεί να είναι εκρεμές και σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Τέταρτος λόγος για τον οποίο εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Ο θεσμικός ρόλος. Πρώτη φορά εμείς μπορούμε σαφώς να πούμε ότι είμαστε κομμάτι της όλης διαδικασίας λήψης απόφασης για αυτές τις αποφάσεις. Εάν με ένα, σε ένα τέτοιο σαφές θέμα αγνοήσουμε ε, τον ε, ρόλο μας, τι θα κάνουμε σε περιπτώσεις άλλων συμφωνιών που δεν είναι τόσο σαφείς όπως τούτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναγνωρίσω ξεκινώντας την προσπάθεια η οποία έχει ήδη γίνει. από πλευρά του εισηγητή μα, Έκανε μια σοβαρή προσπάθεια, μια προσπάθεια θα έλεγα θαραλέα και ταυτόχρονα αποτελεσματική. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής πράγματι τίθενται και ορισμένα θέματα τα οποία αν θέλετε προηγούνται τη σύναψη της συμφωνίας και υπάρχουν και προβλήματα συγκυριακού τύπου για θέματα πιο εξειδικευμένα θα έλεγα και ίσως κάπως πιο δευτερεύοντα. Το θέμα είναι τι γίνεται ακριβώς με τα εδάφη της λεγόμενης Δυτικής Σαχάρας. Ξέρετε ότι στα εδάφη αυτά δεν γίνεται αντικείμενο αναγνώρισης η αρμοδιότητα του ε, Μαρόκου. Υπάρχουν αποφάσεις ομόφωνες οι οποίες δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Μαρόκου. Σχετικά με τους υδάτινους πόρους υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, το Μαρόκο και δεν πρέπει να περιλαμβάνει ε, πιθανότητες αναγνώρισης της κατοχής του εδάφους αυτού από το Μαρόκο για τόσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το θέμα είναι εν πολιτικό. Αλλά από την άλλη εμείς θα πρέπει πράγματι να ασχοληθούμε κυρίως με τα θέματα τα οποία άπτονται της δικής μας αρμοδιότητας. Συνεπώς λοιπόν κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί πιστεύω ότι είναι δύσκολο να γίνει το να δεχτεί κανείς μια συμφωνία τέτοιου τύπου θα έλεγα είναι λήψη πολιτικής θέσης και στην ουσία είναι σαν να κάνουμε ότι αγνοούμε ότι με τον τρόπο που το κάνουμε αναγνωρίζουμε το θεμητό και το νόμιμο της ε, μαροκινής κατοχής. Συνεπώς λοιπόν αναγνωρίζω αυτό το οποίο κάνει ο εισηγητής Μέσω της έκθεσης αυτής ε, εμένουμε σε θέματα τα οποία αφορούν τη συμφωνία χωρίς ε, να αγνοούν πλήρως ε, το ευρύτερο πολιτικό πρόβλημα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με πάρα πολλά ανησυχητικά θέματα τα οποία εμπλέκονται στη συμφωνία αυτή, θέματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. ο εισηγητής ε, έκανε μια πάρα πολύ καλή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει επίσης εδώ και πάρα πολύ καιρό τις βαθύτατες αντιρρήσεις τις οποίες έχουμε. Και με τη συμφωνία αυτή και με το περιεχόμενό της και με τον τρόπο με τον οποίο έχει εφαρμοστεί η προηγούμενη συμφωνία μέχρι τώρα. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν άπτονται των πολιτικών μας θέσεων. Παρ' όλα αυτά είμαστε κατά της αρχής που επιτρέπει την λειτουργία και την ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν σοβαρότατες αντιρρήσεις, αντιρρήσεις όχι μόνο πρακτικές, όχι μόνο ιδεολογικές, αλλά και θεσμικές ουσιαστικά, και αυτά όλα πρέπει να επηρεάσουν τη λήψη θέσεών μας. Πρέπει να υπάρξει αναδιαπραγμάτευση. Και θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο σε μια πρώτη φάση τις αρνητικές επιπτώσεις που μια τέτοια απόφαση αρνητική θα έχει στους αλλιευτικούς τόλους στα ύδατα του Μαρόκου. Η λύση θα πρέπει να περνάει όμως όπως και να έχουν τα πράγματα από την εξαίρεση των υδάτων που ανήκουν στην Δυτική Σαχάρα. Ο λαός των Σαχαραούι έχει εκλεκτούς και αναγνωρισμένους αντιπροσώπους σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει πάντα να μπορούν να εκφραστούν και να μεταφέρουν τις ανησυχίες του λαού τους. Αυτή στιγμή γίνουν σεβαστές οι προϋποθέσεις αυτές, τότε μπορούμε να περάσουμε ίσως σε μια κάποια συμφωνία. Θα πρέπει δηλαδή σε καμία περίπτωση να μην αγνοήσουμε τους νόμιμους εκπροσώπους του λαού της Σαχάρας. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Χάγκλουν για την έκθεσή του, ακόμα και αν δεν συμφωνώ καθόλου με τα συμπεράσματά του. Είναι αλήθεια ότι η γνωμοδότηση εκ των υστέρων η οποία μας δόθηκε ασκεί κριτική έντονη στην συμφωνία αυτή. Τη διάβασα με προσοχή και είναι αλήθεια ότι αυτά που πίστευα από πριν έχουν αλλάξει κάπως. Ε, κάποια θέματα πρέπει να τα συζητήσουμε εκ νέου και με τον Κάρλ Υπάρχουν πάντως αρκετοί λόγοι οι οποίοι με οδηγούν στο να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή αντίθετα από αυτά τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή είμαι ιδιαίτερο ικανοποιημένος που ακούω από πλευρά του Καρλ Άκλουντ ότι πρόκειται για τη συζήτηση μιας αλλιευτικής αλληλείας και όχι ενός διεθνούς γεωστρατηγικού προβλήματος, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση δική μας ευθύνη, ανεξάρτητα από αυτά τα οποία είπε ο Ζωάο και ο Ραούλ προηγουμένως. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Εγώ πήρα πληροφορίες και από τις αρχές του Μαρόκου, οι οποίες με διαβεβαιούν και δεν βλέπω γιατί να μην τις πιστέψω, ότι η βοήθεια που δίδεται κατανέμεται δίκαια σε όλη την ακτή και στην ακτή της Δυτικής Σαχάρα και στις, στους λιμένες του Αγιούν και της Ντάρλα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία, επαναλαμβάνω, η οποία επιτρέπει στις, στα σκάφη με σημαίες κρατών μελών να αλλιεύουν στα ύδατα του Μαρόκου. Είναι μια συμφωνία που έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 27 Φεβρουάριου του 2012, τέσσερις μήνες μένουν δηλαδή. Και σήμερα στην ουσία θα καταγγείλουμε μια συμφωνία η οποία έχει ισχύ περαιτέρω ε, τεσσάρων μηνών. Ε, τώρα αυτό μου φαίνεται λίγο ζημιογόνο. Γιατί αν καταγγείλουμε τη συμφωνία, έχω την αίσθηση ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπραγματευτούμε μια καινούργια συμφωνία με το Μαρόκο. Εγώ θέλω να υπάρξει μια καινούργια συμφωνία με το Μαρόκο, κάτω από άλλες συνθήκες ίσως, κάτω από διαφορετική μορφή ίσως. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να το κάνουμε έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντά μας, το Μαρόκο να σέβεται κάποιους κανόνες τους οποίους εμένουμε και πάρα πολύ σωστά, και νομίζω για μια ακόμη φορά ότι θα ήταν ε, πολύ σοβαρό λάθος και πολύ σοβαρό για το μέλλον να καταγγείλουμε τη συμφωνία αυτή. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά, η συμφωνία αυτή είναι σημαντική για το Μαρόκο, η συμφωνία αυτή είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Κάποιοι εδώ μιλούν μόνο για γεωπολιτική. Όπως σας είπα και όπως σας θυμίζω, το Μαρόκο με πολύ ίσως soft τρόπο αλλά με έξυπνο τρόπο είναι σε μια περίοδο εκδημοκρατισμού όπως και άλλες περιοχές, χώρες μάλλον της περιοχής δεν πρόκειται για μια επανάσταση, πρόκειται για μια μετάλλαξη αν θέλετε του καθεστώτος της χώρας αυτής και νομίζω ότι θα ήταν πολύ αρνητικό το μήνυμα που θα στέλναμε κατά τη συμφωνία. Συνεπώς λοιπόν εγώ θέλω να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή ως έχει. Κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να διαπραγματευτούμε για τα επόμενα χρόνια κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω αυτό το θέμα το συζητάμε εδώ και αρκετούς μήνες. Η έκθεση του κύριου Χάγκλουν που στηρίζεται την αξιολόγηση του αντικτύπου που είχαμε όλη την ευκαιρία να εξετάσουμε. Είναι μια πολύ σοβαρή έκθεση, αυτό αληθεύει. Αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία πιστεύω ότι αντανακλούν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες θέσεις που ακούσαμε να εκφράζονται σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα. Τώρα, στην σελίδα 96, στο θέμα του περιβάλλοντος, λέει ότι η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο επηρεάζει μόνο 4% ε, της αλίες και ε, οι αλλιευτικοί στόλοι Μαρόκου ε, αλλιεύουν μόνο στα δικά τους ύδατα και εδώ όταν ε, αναφέρεται στο στόλο εννοεί και τρίτης χώρας στόλους. Άρα ο πως θα είναι ελάχιστος. Ε, οι στόλοι ευρωπαϊκοί που αλλιεύουν στα ύδατα του Μαρόκου είναι ελάχιστοι. Λέει ότι υπάρχει ευκαιρία για τους στόλους μας να αλλιεύουν σε ε, ξένα ύδατα. Αναφέρεται ε, στην ανάγκη να υπάρξει καλύτερος διάλογος. Και με βάση όλα αυτά τα πολιτικά θέματα και τη συζήτηση που έχουμε ακούσει, ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την παράταση μιας συμφωνίας. Και στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας θα ε, γίνει μια αξιολόγηση των ε, οικονομικών και ε, γεωγραφικών κριτηρίων για να αξιολογηθεί αν είναι επωφελής αυτή η συμφωνία. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, ότι αυτή η παράταση της συμφωνίας στα πλαίσια του σημείου 4 θα περιλαμβάνει και μια έκθεση αξιολόγησης που θα πρέπει να διενεργηθεί δύο μήνες πριν από την εκπνοή αυτής της ε, συμφωνίας ή πριν από την περαιτέρω παράταση της συμφωνίας. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. θα πρέπει να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε επί της διαπραγμάτευσης ενός νέου πρωτοκόλλου που θα περιλαμβάνει τις βελτιώσεις που θέλουμε να δούμε και που περιλαμβάνονται σε αυτή την Επιτροπή και ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτό το έργο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε στην Επιτροπή. Βέβαια θέλουμε να δούμε βελτιώσεις στη συμφωνία και φυσικά δεν θέλουμε να προσυπογράψουμε οποιαδήποτε συμφωνία που να είναι επιβλαβής σε χώρες εταίρους όπως είναι το Μαρόκο και δικούς μας τόλους επίσης. Αλλά ας μην ξεχνούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα και ποια είναι η κατάσταση για τους ίδιους τους αλληλείς. Παρόλο που αυτή η συμφωνία δεν θα έχει σχεδόν καθόλου αντίκτυπο, θα είναι καλύτερο να υπάρχει παρά να μην υπάρχει καμία συμφωνία. Είναι σημαντικό για το Μαρόκο να ευθυγραμμίσει το σύστημά του με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ε, θα πρέπει να αναμένουμε από τις αρχές ε, κάποια πληροφόρηση. Αλλά καταρθώσαμε ε, να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που είχαμε μέχρι στιγμής και αυτά δημοσιεύτηκαν στην έκθεση της αξιολογήσης των αντικτύπων. Εγώ είμαι υπέρ της παράτασης αυτής της συμφωνίας ως πρώτο στάδιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας με το Μαρόκο, αλλά πρέπει να είναι μια τελείως διαφορετική συμφωνία σε σχέση με αυτή που έχουμε τώρα. Πρέπει να είναι καλύτερη από την τωρινή, πρέπει να είναι πολύ πιο υπεύθυνη από την τωρινή. Στους τελευταίους μήνες έχουμε στείλει πολλά μηνύματα προς τους ε, Μαροκινούς ε, και οι Μαροκινοί ε, και μάλλον οι, οι αλληλείς τη της Ευρώπης ήξεραν πώς έχει η κατάσταση. Τελευταία, τους τελευταίους μήνες έχουμε πολλές πολλά δημοκρατικά κινήματα στο Μαρόκο, έχουμε πολλές αλλαγέ που βεβαίως πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μα και δεν πρέπει φυσικά να τι αμφισβητήσουμε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η παράταση έτσι όπω έχει δεν μπορούμε να, την, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ήταν ελεύθερη η ψηφοφορία στην ομάδα μου και ο καθένας ψήφισε ανάλογα με το τι του έλεγε η συνείδησή του. Νομίζω όμως ότι τα μηνύματα που στείλαμε δεν ήταν απόλυτα σαφή. Και επίσης η ψηφοφορία η πρώτη έγινε γιατί, χωρίς να ληφθεί υπόψη από του Κοινοβουλίου. Και ε, τέτοιου είδου μηνύματα θα πρέπει να τα στέλνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλάβουν και οι Μαροκινοί ότι είμαστε σοβαροί και ότι θέλουμε να διαπραγματευτούμε μαζί τους. Έτσι ώστε για να έχουμε μια πολύ καλύτερη από όλες τις συμφωνία και πιο υπεύθυνη. Αυτή τη, αυτή τη φορά νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τα πράγματα από την αρχή και να μην μπούμε στην όλη διαδικασία σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Θέλουμε λοιπόν να στείλουμε τέτοια μηνύματα προς το Μαρόκο. Θέλουμε η επόμενη συμφωνία να είναι πιο υπεύθυνη και ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο η Κομισιόν αλλά και οι Μαροκινοί θα υποχρεωθούν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάκτον. Και κλείνω τον κατάλογο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές που μίλησαν για την αλληλεγγύη με, τους, με τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας. Είναι απαράδεκτο να σκεφτόμαστε, να αγνοήσουμε το πώς έχει η κατάσταση εκεί και να νομιμοποιήσουμε ίσως την, το, τη διαμάχη που υπάρχει για την επικράτεια επιτόπου όπως λέει και το επεξηγηματικό σημείωμα του εισηγητή τα ε, στοιχεία που έχει ο ίδιος δεν ξεκαθαρίζουν καθόλου το σημείο αυτό και είμαι απογοητευμένος που μια μεγάλη πλειοψηφία ε, ευρωβουλευτών φοβούνται να πάνε το θέμα αυτό μέχρι το δικαστήριο. Αλλά πέρα από αυτό, τα χρόνια, όσα χρόνια ακούω εγώ συζητήσει ε, τέτοιε για την αλληλεία και τι συμφωνίε, είμαι όλο και πιο πολύ σκεπτικό για το πόσο αξία έχουν. Έχουμε κάποιε αξιολογήσει βεβαίω, οι οποίε εντάξει είναι λίγο στο όριο του να είναι αντικειμενικέ. Πολλέ φορέ έχουμε δυσκολία να ε, αποδείξουμε την αξία αυτών των συμφωνιών για οποιονδήποτε, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε ούτε καν αυτό. Ο εισηγητή λέει σαφώ ότι η αξιολόγηση λέει ότι το, η συμφωνία δεν έχει τελικά βοηθήσει στην ανάπτυξη του αληφτικού τομέα στο Μαρόκο. Οπότε υπάρχουν ε, επαρκείς λόγοι για να ε, συμφωνήσουμε νομίζω ε, με τον εισηγητή να μην συνεχιστεί η συμφωνία και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να καταψηφίσουμε μια εκ νέου σύναψη τέτοια συμφωνία. Ναι, ευχαριστώ. Να κάνω κι εγώ μια σύντομη παρατήρηση. Όπως είδαμε και στην Ολομέλεια, Είχαμε 301 ε, ψήφους υπέρ και 220 ε, ψήφους κατά και κάποιες αποχές. Αυτά είναι τα ε, αριθμητικά στοιχεία που έχω σημειώσει εγώ. Οπότε πρέπει να δεχτούμε και το αποτέλεσμα της ολομέλειας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό λοιπόν έχει κλείσει, εκτός εάν πρόκειται κάθε μήνα να υποβάλουμε νέα πρόταση συμφωνώ με τα όσα, είπε, τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του κ. Χάκλαν. Ε, και εγώ ήμουνα παρούσα στις διαπραγματεύσεις και μάλιστα ήμουνα από αυτούς που εξέφρασαν ε, πολύ ε, κριτικά σχόλια για την συμφωνία αυτή. Οπότε ξέρω ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε λοιπόν το ζήτημα. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικές συζητήσεις και νομίζω ότι και το Μαρόκο καταλαβαίνει και πιστεύει ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Ο ευρωπαϊκός αλλιευτικός τομέας, ο κλάδος επίσης γνωρίζει ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε στο μέλλον. Το πρωτόκολλο αποτελεί μια παράταση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μπάλωμα που σκέφτηκε η Κομισιόν γιατί δεν μπορεί να λύσει όλα τα θέματα εγκαίρως. Δεν νομίζω όμως Αξίζει την προσοχή μας, αξίζει το χρόνο μας να έχουμε οποιαδήποτε έτσι παρέμβαση σε αυτό. Δεν το νομίζω τουλάχιστον εγώ. Οπότε εγώ προτείνω ο κύριος Χάγκλουντ όταν θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια να ζητήσει μια νομοθετική πρόταση και να θέσουμε σαφώς τις προοπτικές που πρέπει να υπάρχουν για μελλοντικές συμφωνίες με το Μαρόκο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να πούμε όχι. Αν θέλουμε να είμαστε ε, ρεαλιστές και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να υποβάλουμε μία νομοθετική πρόταση η οποία θα μπορούσε να εγκριθεί και να δώσει ένα σαφές μήνυμα για το ποιες θα είναι οι αλληλευτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου. Έτσι όπως τις βλέπουμε εμείς τουλάχιστον. Η Κομισιόν τώρα παρακαλώ. Thank you. Ε, thank you, ε, Mrs. Ε, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Απλά να κάνω κάποιες διευκρινήσεις για τεχνικά θέματα. Τα περισσότερα επιχειρήματα έχουν γίνει και είναι ενθαρρυντικό που ακούσαμε ότι υπάρχει μια βασική βούληση να εξεταστεί μια νέα συμφωνία και ότι δεν υπάρχει βασική ε, αντίθεση σε μια συμφωνία με το Μαρόκο. Ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να δείξω σε σχέση με αυτά που άκουσα και από την Πρόεδρο είναι ότι το θέμα της φορολογίας και της χρήσης ε, των χρημάτων φορολογουμένων είναι παραπλανητικό. Διότι στην ουσία συζητάμε εδώ μια ενός έτους παράταση και αυτή η περίοδος έχει ήδη εκπνεύσει. Ε, και τα χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν ε, ούτως ή άλλως και πρακτικά για τον φορολογούμενο δεν έχει καμία διαφορά εδώ και δεν ε, θα γίνουν περαιτέρω εξοικονομήσεις. Όντως, ε, η έκθεση εξολόγηση λέει ότι οι τεχνικές συνθήκες της συμφωνίας θα πρέπει να διαπραγματευτούν. Αλλά εδώ συζητάμε μία παράταση ενός έτους με όλες τις συνθήκες όσοι είχαν, άρα δεν υπήρχε πιθανότητα να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση. Μια τέτοια τροποποίηση θα έπρεπε, εάν ε, διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους όρους αναφοράς οποιασδήποτε νέας συμφωνίας. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να διορθώσω σχετικά με το πλεόνασμα και την υπερεκμετάλλευση έχει δηλεχθεί από διάφορους ομιλητές αυτό το θέμα, αλλά στη συμφωνία αυτή εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλιεύουμε σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε ένα πολύ μικρό μερίδιο ε, των αλλιεύματων στο Μαρόκο και τα είδη τα οποία ε, τη χάνουν δεν είναι αυτά ε, που βρίσκονται σε αυτή την συμφωνία από πλευράς διατήρησης. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θέτει οποιοδήποτε κίνδυνο. Αφετέρου, αν θέλουμε να έχουμε με το Μαρόκο μια δυνατότητα να επηρεάσουμε την πολιτική και τους ή να τους σωθήσουμε προς περαιτέρω ε, διατήρηση είναι αυτός ο μόνος τρόπος που έχουμε αν θέλουμε να επιδιώξουμε αυτό το στόχο και να ασκήσουμε κάποια, ε, κάποια ε, πίεση στον τρόπο που διαχειρίζονται το στόλο τους ή τον τρόπο που αλλιεύουν και μη μαροκινοί που αλλιεύουν σε αυτά τα ύδατα. Από αυτή την έννοια λοιπόν μια πιθανή νέα συμφωνία μετά από αυτή θα πρόσφερε τη δυνατότητα άσκησης κάποιας επιρροής στο θέμα της συντήρησης. Τα ωφέλη τώρα στο νότιο μέρος της περιοχής. Είχα, πήραμε πληροφόρηση, περιμένουμε και άλλες πληροφορίες για την παράταση του ενός έτους. Οι πληροφορίες θα ε, πρέπει να... Ε, βέβαια ε, δόθηκαν αργά και ελπίζουμε να έχουμε εντός του μηνός επαρκείς νέες πληροφορίες από το Μαρόκο για να εξηγήσουμε αποτελεσματικά ότι έχει αποφεληθεί και ο Νότος και το είπε και ο κύριος Καντέκ ότι οι πληροφορίες που έχουν δοθεί είναι κάπως ενθαρρυντικές. Τέλος, στο θέμα της ε, εάν τερματιστεί αυτή η συμφωνία, ποιε θα είναι οι επιπτώσει, Υπάρχουν δύο συνιστώσει του Ευρωπαϊκού Στόλου που αλλιεύει στην περιοχή. Έχουμε μεγάλε εταιρείε και ο κ. Χάγκλουν ε, μπορεί ε, να αυτές θα μπορούν να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους και να αλλιεύουν κάπου αλλού. Αλλά δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε την ε, επίπτωση και την επίδραση σε περίπου 100 αλλιευτικά σκάφη, τα οποία είναι μικρότερου μεγέθους και τα οποία αλλιεύουν επίσης σε πλαίσια αυτής της συμφωνίας και ίσως να δυσκολευτούν πολύ να μετεκατασταθούν. Ελπίζουμε ότι αυτή η παράταση ενός έτους θα εγκριθεί και ότι θα την ε, εγκρίνεται και είναι σαφές ότι αυτό θα ανοίξει το δρόμο για μια πιθανή επαναδιαπραγμάτευση μιας μελλοντικής συμφωνίας. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει υπό διαφορετικούς όρους ε, με μια επαναδιαπραγμάτευση των τεχνικών παραμέτρων που θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις αλληλευτικές ε, ευκαιρίες. Ευχαριστώ κύριε Χάγκλου. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εδώ και δύο χρόνια ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα μαζί σας και είπαμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και μας είπατε ακριβώς αυτά τα οποία μας είπατε και τότε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις αλλά όχι να ξεκινήσουμε αυτή τη στιγμή άλλες διαπραγματεύσεις. Η εμπιστοσύνη μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό είναι περιορισμένη. Εσείς επαναλάβατε αυτό που μας είπατε και πριν δύο χρόνια, δυστυχώς. Εγώ, κοιτάξτε, δεν θέλω να σώσω μόνο τα χρήματα των ε, φορολογουμένων. Δεν είναι απλά για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Προφανώς και οι Μαροκινοί θα πρέπει να πληρωθούν για φέτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι σαφές. Το θέμα είναι αν θέλουμε εμείς να ευλογήσουμε κακές δαπάνες από εδώ και πέρα. Είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου ε, μάλλον Προϋπολογισμών και μπορώ να εξοικονομήσω χρήματα πολύ περισσότερα σε άλλους τομείς. Δεν είναι αυτό που θέλω. Τώρα για το περιβάλλον. Το θέμα είναι να δούμε αν συμφωνούμε ή όχι με την υπεραλίευση. Υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα από ότι εκεί. Το θέμα είναι όμως αν εμείς θα δεχθούμε πολιτικά την υπεραλίευση και μου κάνει εντύπωση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πολιτικές ευθύνες, πρέπει να αναλάβετε και εσείς τις δικές σας, λέει, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την επικοδομητική τους συνεισφορά. Θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό Ξέρουμε ότι το πρόβλημα ιδιαίτερα σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα είναι ακαθόδες. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συζήτησης αναλώθηκε λοιπόν για τη Δυτική Σαχάρα. Είναι ένα θέμα το οποίο για πολλούς από εσά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας, η συμφωνία αυτή θα ήταν πάρα πολύ προβληματική. Αυτό μας το ξεκαθάρισε η νομική υπηρεσία. Διάβασα και άλλες νομικές αξιολογήσεις Υπεψήφισα τη συμφωνία αυτή και ο λόγος ήταν γιατί πιστεύω ότι θα ήταν καλό για όλες τις πλευρές και το Μαρόκο να διευκρινίσουν καλύτερα την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς κάνοντας το αυτό, αφού το έκανα, διάβασα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και στο γραφείο μου πολλές νομοδοτήσεις, νομικές, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί νομομαθείς οι οποίοι καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα πλέον. Τώρα σχετικά με αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Και για όσους είπατε ότι δεν διαφωνείτε μαζί μου, Κατανοώ αυτά τα οποία άκουσα. Κατανοώ τις ανησυχίες που έχουν ορισμένοι από εσά για τους αλληλείς, τους εργαζόμενους γενικά και τους μικρούς τόλους. Αυτό είναι ένα επιχείρημα, ίσως το μόνο καλό επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, αλλά αν το ζυγίσει κανείς, το σταθμίσει σε σχέση με τα αρνητικά επιχειρήματα, δεν είναι πολύ ισχυρό σαν επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Τώρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Μαρόκο, αυτά που γίνονται είναι θετικά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μας απασχολεί στη συγκεκριμένη φάση, δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη έκθεση. Ας μην το αγνοήσουμε λοιπόν, το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και όχι εμείς. Είναι θέμα στάσης. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μικρός ο χρόνος που μένει, οπότε πρέπει να πούμε ναι. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι είναι παραδειγματικό και πρέπει να πούμε όχι. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσουμε θα πρέπει εμείς να δούμε αν θέλουμε εμείς να ευλογήσουμε πολιτικά ένα πρόγραμμα το οποίο και οικονομικά και οικολογικά δεν είναι υποστηρίξιμο. Εγώ δεν ήθελα να ξοδέψω πάρα πολύ χρόνο σε θέματα απόλυτα αρνητικά. Νιώθω μια κάποια δυσθυμία γιατί είναι δύσκολο πολύ το θέμα αυτό. Δεν ήθελα να ξεκινήσω με θέματα δυσάρεστα σήμερα το πρωί γιατί ήδη όταν το έχουμε κάνει χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό λίγο καλύτερα θα ήταν πολύ πιο εύκολη η κατάσταση για όλους. Είχαμε μια ιδιαίτερα επικοδομητική συζήτηση με τους Μαροκινούς και λυπάμαι για τους Μαροκινούς γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν το θέμα. Ήταν πολύ πιο εύκολο να συνεργαστεί κανείς και με τις αρχές του Μαρόκου παρά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Τέλος, Χαίρομαι γιατί συμφωνούμε όλοι ε, λέγοντας ότι το Φεβρουάριο έχουμε ανάγκη από μια καλύτερη συμφωνία. Δεν ξέρω ποιε θα είναι οι πλειοψηφίε γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να ψηφίσουμε. Διάφοροι βουλευτές για διαφορετικούς λόγους έχουν διαφορετικές απόψεις αλλά παρόλα αυτά ένα πάνω στο οποίο συμφωνούμε είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια καλύτερη νομοθετική πρόταση ανεκτή τεχνικά Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε ε, θετικό μήνυμα, δεν μπορούμε να αναλάβουμε μια τέτοια πολιτική ευθύνη. Ταυτόχρονα όμως αυτό το οποίο πρέπει να δείξουμε προς τους Μαροκινούς είναι ότι θέλουμε αλλαγές. Και θυμίζω, το βασικό είναι ότι πριν δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυριζόταν αυτά τα οποία συνεχίζει να ισχυρίζεται και σήμερα και αυτό μας απογοητεύει τα μάλα δεν μπορούμε να ακούμε τα πράγματα να μην αλλάζουν με τέτοιο τρόπο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος μας είπε τα ίδια που μας είχε πει ένας άλλος κύριος πριν δύο χρόνια ε, και ε, εν τω μεταξύ είχε έρθει και μια συμπαθεστάτη κυρία η οποία μας είπε και αυτή τα ίδια προβλήματα, τα ίδια θέματα και την ίδια λογική. Λοιπόν δεν αλλάζει η στάση μου απέναντι σε αυτό. Σας είπα ποια είναι η άποψή μου και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί τώρα να δούμε σε τι πλαίσιο θέλουμε να κινηθούμε για τη νέα συμφωνία. Και να μας εξηγήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποια πεδία πιστεύει ότι μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος. Όπως έχω πει, δεν είναι ότι δεν θέλουμε συμφωνία, αλλά θέλουμε καλύτερη συμφωνία. να σας αναφέρω λίγο το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 22-23 Νοέμβρη. Ολομέλεια, ψηφοφορία στην Ολομέλεια, είτε τον Δεκέμβρη είτε τον Ιανουάριο. Θα έχει δουλειά βόλικη ο συγκητής μας. Πάμε στο σημείο 3α που είναι το νέο πρωτοκολλό με την Βουινέα ε, Μπισάου. Κύριε Χάγκλιν, θέλετε να, δώσετε, πάρετε το λόγο τώρα, θέλετε να μιλήσει πρώτα η Επιτροπή. Όχι, ωραία, να εξηγήσω γιατί το βάλαμε στην ημερήσια διάταξη και θα, το, θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Ε, προσπαθούμε εδώ να συνεργαστούμε καλύτερα με την Κομισιόν για όλες τις διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ε, Έχουμε καιρό που ξεκίνησαμε τι διαπραγματεύσει για το θέμα αυτό, αλλά έχουν μείνει λίγο πίσω σε ό,τι αφορά την όλη διαδικασία ε, έγκριση. Οπότε θέλουμε να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Όπω και με το Μαρόκο. Αν κάνουμε λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων σήμερα, θα μπορούσαμε να υποβάλουμε στην επόμενη συνεδρίαση την έκθεση, οπότε θα ληφθεί πιο γρήγορα η απόφαση. Οπότε γι' αυτό, για λόγους δηλαδή χρονοδιαγράμματος, θέλαμε να κάνουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Και βεβαίως να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Μετά, αφού μιλήσει η Κομισιόν, θα μιλήσω και εγώ πάλι. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, παρακαλώ. Αυτή η συμφωνία με την ε, Γουνία Μπισάου πάλι περιλαμβάνει μία ετήσια παράταση. για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι αλληλευτικές δραστηριότητε. Η συμφωνία ε, διακόπηκε λόγω κάποιων ε, θεμάτων με ανθρώπινα δικαιώματα και συμφωνήσαμε με την Γουινέα Μπισάου να συνεχίσουμε για ένα χρόνο, με ένα χρόνο παράταση δηλαδή, και με μία ρήτρα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην ε, συμφωνία. Οπότε, ίδιες οι συνθήκες όπως, οι προηγούμενοι, όπως τις προηγούμενες ε, συμφωνίες. Παράταση λοιπόν για ένα χρόνο και σε ένα χρόνο θα ε, διαπραγματευτούμε μια νέα συμφωνία η οποία διαρθρωτικά θα είναι καλύτερη. Το πρωτόκολλο αυτό εφαρμόζεται από τις 16 Ιουνίου και εκπνέει 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Εν τω μεταξύ, θέλουμε να, διατηρηθεί, να διατηρηθούν οι ελευτικές ευκαιρίες και να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξουν περαιτέρω συμφωνίες μετά από το επόμενο έτος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάγκλουντ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, η συμφωνία αυτή είναι όντω καλύτερη από την ε, προηγούμενη εταιρική συμφωνία που είχαμε ε, συζητήσει. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν που συμπεριέλαβε το, τη ρήτρα αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί χωρί αυτό Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για μας να συμφωνήσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι κάθε άλλο παρακαλή. Βεβαίως μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό και, στην, και σε σχέση με αυτά που είπαμε πιο πριν για το Μαρόκο, ότι όντως πρέπει να τα συζητήσουμε πολύ καλά τα θέματα αυτά, όπου όταν αποφασίζουμε να μην δίνουμε συγκατάθεση λόγω πολιτικών καταστάσεων. Άλλοι συνάδελφοι βέβαια είπαν ότι θα πρέπει να δούμε μόνο τα ληφτικά θέματα και την πολιτική ευθύνη θα πρέπει να την αναλάβουν άλλοι. Είναι δύσκολη η εξέβρεση ισορροπίας, αλλά σε σχέση με τα αληφτικά θέματα θα πρέπει να δούμε και την αξιολόγηση εξ post, την εκ των υστέρων που προέκυψε από την Κομισιόν, η οποία λέει ότι είναι καλή η συμφωνία αυτή, είναι ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές και η, συμβολή της, η οικονομική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική για τη Γουνέα Είναι πολύ φτωχό το κράτος αυτό. Οπότε είναι καλό που μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο συμβάλλοντας οικονομικά. Σε σχέση με το Μαρόκο δηλαδή, το Μαρόκο είναι οικονομικά δυνατό, ε, και τα οικονομικά ωφέλη για τους Μαροκινούς δεν είναι τόσο σημαντικά για την, από, τη, από τη συμφωνία μας, αλλά για την Γινέα Μπισάου νομίζω ότι όντω είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία και νομίζω ότι θα πρέπει όντως να είμαστε και εμείς θετικοί προς την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα όμως και η Κομισιόν να δει λίγο περισσότερο το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι συμβαίνουν διάφορα ε, ε, γεγονότα που τα ακούμε στα ΜΜΕ. Αν μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο το τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς σκοπεύετε να το παρακολουθήσετε, να μην υπάρχει δηλαδή μια απλή δήλωση, αλλά να μπορούμε με κάποιο τρόπο να επηρεάσουμε τα πράγματα. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, θα μας κάνετε μεγάλη χάρη για να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας και να διαβάσουμε βεβαίως λίγο πιο ε, σε βάθος την έκθεση. Ευχαριστώ. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεση θα παρουσιαστεί στην συνεδρία του Νοέμβρη. Ως τότε θα μελετήσουμε την πρόταση της Κομισιόν πολύ προσεκτικά. Ευχαριστούμε κύριε Χάγκλον. Πάμε στο επίομενο σημείο, σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Ε, πολιετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα έχει το λόγο και θα δώσουμε το λόγο και στην Κομισιόν. Η απόφαση έχει ληφθεί από πέρσι ήδη από την ΆΙΚΑΠ στο Παρίσι. Κύριε Ρωμέδα, έχετε το λόγο. Ε, και τι Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία αν θέλετε έχει δύο πλευρές. Από τη μία υπάρχει το τεχνικό κομμάτι ένα τεχνικό κομμάτι το οποίο μας υποχρεεί σαν ευρωπαϊκό όργανο να διεθνοποιήσουμε αν θέλετε την αντιμετώπιση του προβλήματος και της απόφασης η οποία είχε γίνει δεκτή. Και από την άλλη υπάρχει μια συζήτηση ενδοευρωπαϊκή που αφορά τη διαχείριση του αλλιευτικού, του αλλιευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξέρετε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν εδώ να αντιμετωπίσουμε το θέμα το οποίο θα μας επιτρέψει ε, στις συμφωνίες που έχουν γίνει δεκτοί στα πλαίσια της ΕΚΑΤ να, να γίνουν πραγματικότητα, να ισχύσουν εν πάση περιπτώσει, χωρίς σε καμία περίπτωση ε, να ξεπεράσουμε τα ελάχιστα τα οποία προτείνει η συμφωνία αυτή. Τι εννοώ με αυτό. Αυτά που υιοθετήσαμε στα πλαίσια των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, η ICAT, pero que en algunos Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να κάνουμε δεκτά αυτά τα οποία λέγει τα Ταλικάτα. Από την άλλη, αν η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το δέχεται, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα στα πλαίσια των προτάσεων την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά πρώτον, γι' αυτό δεν είναι καθόλου θα έλεγα. Δευτερεύον είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται με τη βιομάζα η οποία ανταποκρίνεται στη μέγιστη αηφόρο απόδοση η οποία θα πρέπει να είναι σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 60%. Αυτό το 60% δεν μας εμποδίζει σε καμία περίπτωση να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι μια λογική θα έλεγα απόφαση. Νομίζω ότι το 100% είναι ε, κάτι το οποίο δεν μπορεί να στηριχθεί απόλυτα. Νομίζω ότι η κατάσταση απαιτεί να δοθεί μία απάντηση. Η απάντηση αυτή θα πρέπει να είναι πιστική. Η συμφωνία η ΚΑΤ έτσι και αλλιώ προτείνει 60%. Γιατί να περάσουμε θα πούν ορισμένοι μονομερός πέραν του 60%. Εδώ θα απαντήσω λέγοντας ότι αν πράγματι εμείς θέλουμε και μπορούμε να εκπληρώσουμε τον συγκεκριμένο στόχο, είναι σαφές ότι θα πρέπει να περάσουμε σε διαδοχικές φάσεις αντιστάθμισης, γιατί θα έχουμε ξεπεράσει τα όρια και τις προθεσμίες. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι στο παρελθόν εμείς θέσαμε αυτούς όρια τα οποία σχεδόν πάντα ξεπεράσαμε. Δεν σεβαστήκαμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο αυστηροί και πιο πειθαρχημένοι σε σχέση με τον καθορισμό των ορίων και ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο θαραλέοι σχετικά με τους στόχους τους οποίους έχουμε για την αποκατάσταση της ισορροπίας των αλλιευμάτων και σχετικά με την μέγιστη αηφόρο απόδοση που είναι ο βασικός στόχος των προτάσεων της ΛΕΚΑΤ και που θα πρέπει να μεταφερθεί σε κάποια φάση στο κοινοτικό δίκαιο. Υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση της προβληματικής αυτής, είναι η νομική διάσταση. Δεν μπορούμε να υιοθετούμε αποφάσεις οι οποίες να είναι ασύμβατες με το νομοθετικό πλαίσιο. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι περιοριστικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα των αποφάσεων της ΔΕΚΑΤ έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και στο εσωτερικό της και εκτός. Κάποιοι από εμά πήραμε ε, μέρος στις συναντήσεις αυτές ε, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας και στο Παρίσι και αυτό δείχνει την ανάγκη που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει θέσει, οι οποίε να είναι συμβατέ με το υπάρχον νομικό πλαίσιο όπω ακριβώ προβλέπεται ε, στο άρθρο 7. Πρέπει να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες ήδη περιλαμβάνονται στην οδηγία πλαίσιο. Αυτά όλα μας υποχρεώνουν τελικά και εμένω σε αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μας επιβάλλεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος μέσω της τροπολογίας της. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια αναθεώρηση και είναι κάτι το οποίο συνδέεται με μια αναφορά στο 70% ανάκτησης της βιομάζας. Ακριβώς αυτό είναι το οποίο απαιτείται να γίνει πριν από κάποια προθεσμία ή πριν κάποια συγκεκριμένη περίοδο. Νομίζω ότι κάποιες από τις τροπολογίες που έχει καταθέσει η συγκεκριμένη επιτροπή το επιδιώκουν αυτό, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι αυτά τα οποία υιοθετούμε εμείς εδώ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι ασύμβατα με την οδηγία πλαίσιο. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο και το οποίο προέρχεται και αυτό από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ένα τρίτο στοιχείο λοιπόν, το οποίο θα πρέπει να επιδιωχθεί είναι ό,τι έχει σχέση με την ανάκτηση των ποσοτήτων. Από την άλλη υπάρχει το μέγεθος των κλοβών. Αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ σχετικά με το μέγεθος των κλοβών είναι ότι τα μέσα, οι κλοβοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται εκτός των δικαιοδοσιών των συμβαλωμένων μερών θα πρέπει και αυτοί να ανήκουν τα πλαίσια, να εντάσσονται στα πλαίσια της ευθύνη αυτών οι οποίοι ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Από την άλλη, οι περιοχές οι οποίες είναι προστατευόμενες και οι οποίες είναι περιοχές καταφύγια που συνδέονται με την αναπαραγωγή και οι οποίες καθορίζονται επίσης σαν προστατευόμενες ζώνες που θα επιτρέψουν την ανάκτηση των ποσοτήτων των αλλιευμάτων είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί επανειλημμένα αλλά το οποίο δεν έχει επιτευχθεί νομίζω συνολικά μέχρι τώρα και είναι το θέμα των καταφυγίων, των αλλιευτικών καταφυγίων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ε, μπει, αν θέλετε, στην τελική του διατύπωση. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο εμείς ε, στην ουσία ε, επιβάλλουμε και πρόστιμα για τον μη σεβασμό κάποιων κανόνων. Υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος συμπεριφορών οι οποίες είναι απαράδεκτες και δυστυχώς τα μέτρα και οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται δεν είναι επαρκώς αποτρεπτικά έτσι ώστε να, να επιτρέψουν την προσφυγή στην χρήση τέτοιου είδους πρακτικών. Θα πρέπει λοιπόν να αυστηριοποιηθούν οι πρακτικές αυτές, οι κυρώσεις αυτές. Στα πλαίσια λοιπόν της ΔΕΚΑΤ μπορούμε να απαιτήσουμε είτε στη δήλωση εκμετάλλευσης, είτε στην κατάθεση η οποία θα γίνει δεκτή στα πλαίσια της επόμενης συνάντησης στα μέσα Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη, να απαιτήσουμε έτσι ώστε η ΝΙΚΑΤ να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή θα έλεγα στάση σε σχέση με τις κυρώσεις εις βάρος αυτών των απαράδεκτων και μη νόμιμων πρακτικών έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και να ε, είναι λειτουργικά. Ένα άλλο θέμα το οποίο δημιουργεί κάποια προβλήματα και το οποίο θα πρέπει όμως ε, να το αντιμετωπίσουμε με τον πιο σοβαρό τρόπο είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες ζώνες στον τομέα αυτό ή κάποιων δραστηριοτήτων θυγατρικών αν θέλετε που επηρεάζουν αρνητικά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Υπάρχουν ορισμένες πρακτικές των οποίων οι συνέπειες είναι θα έλεγα τεράστιες και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες. Ενώ υπάρχουν άλλες πρακτικές και άλλες δραστηριότητες οι οποίες δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα το περιβάλλον. Επαναλαμβάνω, λέει ο κ. Ζωμεβά, υπάρχουν πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να απαγορευτούν. και είναι απαραίτητο να σταματήσουν ορισμένου τέτοιου είδους δραστηριότητες. Εάν πράγματι κάποιες δρακόντιες αποφάσεις δεν ληφθούν τώρα, τότε τα σχέδια που έχουμε για την ανάκτηση των αλλιευμάτων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν, δεν θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα και δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ελαττώσουμε το επίπεδο αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών μας. Περιμένω λοιπόν από τους συναδέλφους τις θέσεις τους. Υπάρχουν λίγες μέρες ακόμα για να συζητήσουμε για τις πιθανές τροπολογίες και νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο προτείνεται εφόσον δεν υπάρχει αμφιβολία είναι το εξής. Κατάθεση τροπολογιών προβλέπεται μέχρι την 24η Νοεμβρίου. Δεν με διορθώνει η Πρόεδρος και η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή στις 19 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον μήνα Ιανουάριο του 12. Έχουμε λοιπόν επαρκέστατο χρόνο για να δουλέψουμε σωστά και νομίζω ότι η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τερματίζεται στις 20 Νοεμβρίου, είναι εύθετη χρονικά και θα μπορέσουμε στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου να έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε στην Κωνσταντινούπολη οι θέσεις μας να ακουστούν γιατί επαναλαμβάνω ότι ο ερυθρός τόνος δεν είναι το κεντρικό θέμα των συνεδριάσεων της ΛΕΚΑΤ. Λοιπόν αυτά και για το χρονισμό του θέματος αυτού, εκτός αν έχουν υπάρξει κάποιες τελευταίες αλλαγές. Δεν έχει κανεί ζητήσει το λόγο, αλλά έχω εγώ κάποια σχόλια που θέλω να κάνω. Το πιο εκπληκτικό είναι το άρθρο 1 που αναφέρεται στην βιομάζα και την πιθανότητα επίτευξης τουλάχιστον ανάκτηση 60%. Αυτό είναι στη σύσταση, αλλά τι γίνεται αν θέλουμε να πάμε πέρα από το 60%. Εμένα με δεν, με ενοχλεί, αλλά το γνώση είναι ότι έχουμε μία βιομάζα, έναν αριθμό και η Podicat έχει έχει θέσει αυτό το επίπεδο. Αν θέσει ψηλότερο επίπεδο, τότε τα άλλα συμβαλόμενα μέρη θα συνεχίσουν να τηρούν την ε, πρόταση. Δεν ξέρω, δεν βλέπω τι ακριβώς κερδίζουμε. Συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τις δυνατότητές τους, αλλά δεν κατανοώ το σημείο σχετικά με τη βιομάζα. Νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της ΕΚΑΤ και να το διατηρήσουμε και στο έγγραφό μας. Διότι υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά συμβαλόμενα μέρη που αλλιεύουν αυτή τη βιομάζα. Ίσως αυτή να ήταν μια καλή εισήγηση για την επόμενη ολομέλεια της ΕΚΑΤ, την επόμενη φορά που θα γίνει η αναθεώρηση της, ε, του επίπεδου πιθανότητων, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην πρόταση της Κομισιόν τώρα. Ε, καταρχήν, λοιπόν, δεν είμαι υπέρ αυτής της τροπολογίας, δεν βλέπω ότι πετυχαίνουμε κάτι με αυτό. Κατά τα υπόλοιπα της πρότασης ε, δεν έχω οποιαδήποτε δυσκολία. ποιε από τις τροπολογίες της Επιτροπής Περιλαμβάνοντος είναι κάπως τρελές πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ε, περί τίνος πρόκειται. Ε, στο θέμα των καταφυγίων, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί εντός της ΕΚΑΤ δεν είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή Περιβάλλοντος μπορεί να ε, θέλει να ενσωματώσει σε αυτό το επίπεδο. Τα καταφύγια είναι πολύ καλά, αλλά νομίζω δεν ε, πρέπει να το δούμε εμείς ε, με πρόταση στην έκθεσή μας. Ε, δεν είμαι εξοικειωμένη με όλες τις προτάσεις, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που τις προτείνουν ε, δεν είναι εξοικειωμένοι και με τις ε, πραγματικότητες, την πραγματικότητα επιτόπου. Ε, όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος της πρότασης, θα δω αυτά που είπαμε και το περασμένο χρόνο και αυτά που συμφωνήσαμε πέρσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια μπορεί να έχει σκληρότερους στόχους, αλλά μόνο αν είναι εφικτή. Και δεν είμαι βέβαια ε, αν μπορούμε να πετύχουμε πολλά με τι τις προτάσεις. Ζεπίπα, από την Κομισιόν. Εκτός μικροφώνου. Όχι, μάλλον ο κύριος Ντονατέλο, εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμείς παρακολουθήσαμε προσεκτικά τις εργασίες σας και στο εσωτερικό αυτής της Επιτροπής, συζητήσεις που έγιναν, αλλά συζητήσει και την ψηφοφορία στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είναι συζητήσεις τις οποίες έχουμε κάνει και στο παρελθόν και θα ήθελα να κάνω κάποιες επιπλέον διαφημίσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που εσείς κάνατε και να μου επιτρέψετε να τοποθετήσω σε διαφορετικό πλαίσιο την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα σχετικά με την μεταφορά του προγράμματος ανάκτησης όπως ακριβώς ε, υιοθετήθησαν το 2010. Καταρχάς και το θυμήσατε εσείς ο ίδιος βρισκόμαστε τώρα σε ένα αυστηρό πλαίσιο μεταφοράς νομοθεσίας. Αυτή η μεταφορά νομοθεσίας είναι βασική για μας και μας διασφαλίζει έτσι ώστε σε επίπεδο εφαρμογής από τα κράτη-μέλη και από τους εμπλεκομένους να έχουμε στη διάθεσή μας, να έχουν όλοι στη διάθεσή τους όλα τα νομικά μέσα τα οποία να μας επιτρέψουν να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε στα πλαίσια της ΛΙΚΑΤ. Η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι να περιοριστούμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και γι' αυτό ορισμένε σκέψεις τις οποίες δεν θα ήθελα να κρίνω δεν μπορούν να γίνουν δεκτές στην πρόταση, στο εσωτερικό της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανεξαρτήτως της σημασίας αν θέλετε και της αξίας τους. Θα ήθελα να το πω αυτό διότι αν μπορεί να φανεί ε, περιορισμένο το κείμενο το οποίο έχετε μπροστά σας είναι όμως ένα κείμενο το οποίο μας εξασφαλίζει ότι εφαρμόζουμε πλήρως και το ταχύτερο δυνατόν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει, υποχρεώσεις οι οποίες θα αναλυθούν από την ΛΙΚΑΤ στο σύνολό της στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, σχετικά περιορισμένο βέβαια, ένα πλαίσιο όμως απαραίτητο έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργούμε απόλυτα συμβατά με τις συστάσεις τις οποίες εσείς οι εκδώσατε. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να θίξω μετά από αυτά που είπε ο εισηγητής είναι ότι σε ορισμένε περιπτώσεις μπορεί να φανεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο από το κείμενο της ΛΚΑ το 2010. Η ιδιαίτερη ισχύει για την αναφορά η οποία έγινε για τους ορισμούς σχετικά με την θέση σε κλωβούς. Να πω ότι ο ορισμός αυτός δεν έχει τροποποιηθεί σε σχέση με την αρχική πρόταση. Απλά αλλάξαμε το κείμενο μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στο άρθρο το οποίο προβλέπει τους ορισμούς ακριβώς το κείμενο το οποίο είχε γίνει δεκτό από την ΛΕΚΑΤ. Μπορούμε να το διευκρινίσουμε αυτό σε διμερές επίπεδο αν θέλετε με όσους ενδιαφέρονται, αλλά η συζήτηση αυτή έχει ήδη γίνει στο παρελθόν στα πλαίσια της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ένα τελευταίο σημείο αφορά την ανάγκη η οποία υπάρχει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαιτούμενα μέσα όχι μόνο για να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι και οι κυρώσεις πιθανώς οι οποίες θα ληφθούν από πλευρά των κρατών μελών να είναι ανάλογες με τις παραβιάσεις, τις παραβάσεις συγγνώμη. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται φυσικά σε αυτού στην πρόταση μεταφοράς, Αυτά είναι στοιχεία δικαίου τα οποία ενυπάρχουν στην υπόλοιπη κοινοτική νομοθεσία. Δεν θεωρήσαμε χρήσιμο σε αυτή τη φάση ε, για να είμαστε ακριβώς συμβατοί ε, με το κείμενο της ΙΚΑΤ να επανισάγουμε συμπληρωματικά μέτρα ελέγχου και συμπληρωματικά μέτρα κυρωτικά των ελέγχων. Αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά λοιπόν τον εισηγητή για μια ξεκάθαρη ανάλυση την οποία έκανε γύρω από τα θέματα που τέθηκαν. Φυσικά είμαστε πάντα στη διάθεσή του για να δώσουμε περαιτέρω απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Ντονατέλο. Κύριο Βαμέβα για να κλείσει η συζήτηση. Αλλάζουμε απόψεις. Έχουμε χρόνο να ολοκληρώσουμε το Έχουμε αρκετό χρόνο να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Έχουμε μια συνάντηση της ΕΚΑΤ στην Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να γερθούν όλα αυτά τα θέματα, παρόλο που δεν έχουμε λύσει όλα τα ζητήματα. Θα βοηθήσει αυτό τη δουλειά της Κομισιόν με τα άλλα συμβαλόμενα μέρη και τη ΆΕΚΑΤ. Νομίζω είναι χρήσιμο για το Κοινοβούλιο να έχει μια σαφή θέση. Υπάρχουν κάποια θέματα που πιστεύουμε είναι σημαντικά. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και θέλουμε να είμαστε σαφείς ως προς ε, την θέση που υποστηρίζει η Κομισιόν εντός της ICAT. Είμαστε ένα από τα κύρια συμβαλόμενα μέρη. Γι' αυτό οι δεσμεύσει μας θα πρέπει να είναι σημαντικές, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης. Ε, θα κλείσουμε εδώ και τώρα τις συζητήσεις στο θέμα αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις τις ερχόμενες εβδομάδες. Θα συνεχίσουμε και το έργο μας. Θα συνεχίσουμε να έχουμε ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας και ελπίζω να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Όπως ε, ακούσαμε, ακούσαμε το χρονοδιάγραμμα, δεν θα το επαναλάβω. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρία. Στο πέμπτο θέμα είναι το θέμα της κυρίας Στράουτμαν, το οποίο αναβλήθηκε στην αυριανή συνεδρίαση. Συνεχίζουμε λοιπόν με το, ε, τα αποθέματα Σολομού της Βαλτικής, αλλά δεν έχουμε εισηγητή ακόμα για το θέμα αυτό. Και δεν τα πάμε πολύ καλά με το χρόνο μας σήμερα και έχουμε και συνεδρίαση και κλεισμένη των θυρών. Γι' αυτό εισηγούμε να αφήσουμε πίσω αυτό το θέμα και να περάσουμε στην έκθεση Φερέιρα σχετικά με την ε, τροποποίηση του κανονισμού 1198 του 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Μήπως ο κύριος Φερέιρα είναι εντός της αιθούσης? Σε αυτή την περίπτωση περνάμε στο επόμενο σημείο. Η ε, κυρία Ρόσμπαχ είναι εδώ. Κυρία Ρόσμπαχ. Όχι. Ναι, είναι εδώ, είναι παρούσα. Κυρία Ρόσμπαχ. Δεν έχω ζητήσει το λόγο. Ξέρω ότι δεν έχετε ζητήσει το λόγο, αλλά έχουμε περάσει στο σημείο 8 που είναι το δικό σας σημείο και είστε η εισηγήτρια του θέματο. Γι' αυτό εγώ σας δίνω την ευκαιρία να πάρετε το λόγο. Παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό εδώ μέσα. Απλά έχουμε πεταχτεί κατευθείαν στο 8. Αν θέλετε να μιλήσετε, αλλιώς μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Έχετε το λόγο λοιπόν. Χαίρομαι που μου δίνετε το λόγο. Ευχαρίστω λοιπόν από δύο λόγια. Πολύ σύντομη είναι η έκθεση. Όπως και σε άλλες περιστάσεις έχουμε δει ότι στη Μεσόγειο αλλά και στη Βαλτική πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα αλληλευτικά μας αποθέματα να παραμείνουν βιώσιμα. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας να συζητήσουμε εντελεχώς το θέμα αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε τα βασικά μας αποθέματα να διατηρηθούν. Μπορεί, ε, κυρία Πρόεδρε, εσείς να μην συμφωνήσατε με τις ε, τροπολογίες που είχαν ε, υποβληθεί για την προηγούμενη έκθεση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αλλά νομίζω ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε το θέμα αυτό. Μιλούμε για ε, βιοτόπους. Ε, ε εντάξει, τώρα τα γερμανικά δεν είναι και η μητρική μου γλώσσα, αλλά νομίζω είναι η γλώσσα που μιλάω καλύτερα αλλά δυστυχώ τη μητρική μου δεν μπορώ να τη μιλήσω σήμερα. Εν πάση περιπτώσει. Κάποια λοιπόν από τα σημεία τα οποία δεν σας βρίσκουν σύμφωνοι ή τέλος πάντων δεν α, συμφωνείτε με αυτά, δυστυχώς θα πρέπει να παραμείνουν στην έκθεση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Μεσόγειο. Θα ήθελα όμως να ακούσω πρώτα την Κομισιόν και μετά, αν χρειαστεί, θα επανέλθω. Ευχαριστώ. Ωραία. Αν δεν σας πειράζει, θα ήθελα κι εγώ να μιλήσω. Ξέρω περί τίνος πρόκειται όταν μιλούμε για τη Μεσόγειο. Δεν μιλούμε μόνο για μεθόδους προστασίας αλλά και για αλλαγή των, των διαδικασιών επιτροπολογία. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Γι' αυτό θέλουμε να συμμορφωθεί και ο κανονισμός με το πλαίσιο που υπάρχει στα πλαίσια της συνθήκη της Λισαβόνα. Συμφωνώ και με την Κομισιόν. Σε πολλά σημεία, αλλά υπάρχουν και κάποια σημεία με τα οποία διαφωνώ. Ας πούμε, σημείο 3 και σημείο 5 Εκεί νομίζω ότι οι αλλαγές για τα παραρτήματα δεν μπορούν να γίνουν μέσω ε, πράξεων και το, σημείο, το άρθρο 3.3 και πάλι δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή τη διαδικασία που προτείνεται για την ε, εξουσιοδότηση. Όπου λοιπόν αναφέρονται πράξεις κατά δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ίσως βέβαια η Κομισιόν θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ευέλικτη για τα σημεία αυτά. Ε, μιλά για ελάχιστα μεγέθη. Ε, σίγουρα οι συνάδελφοι, οι Μεσόγειοι, οι Μεσόγειοι θα ε, συμφωνήσουν ε, ότι θα πρέπει όντω ε, να το δούμε πιο προσεκτικά αν μπορεί η Κομισιόν να ρυθμίζει όλα αυτά τα θέματα μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις πράξεις εξουσιοδότηση. Για όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ. Είναι σημαντικό λοιπόν η Κομισιόν να παρουσιάσει επιστημονικές μελέτες και να λάβει αποφάσεις με βάση αυτά τα επιστημονικά δεδομένα. Αλλά Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι βελτιωμένη η πρόταση αυτή από το τι συμβαίνει τελικά και τι γίνεται σήμερα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία όντως θα πρέπει να τα συμφωνήσουμε, να λαμβάνονται δηλαδή οι αποφάσεις εκεί μέσω ε, κατοξιοδότηση πράξεων. Αλλά ίσως αυτό να μην είναι τόσο σημαντικό. Αλλά για τα παραρτήματα δεν μπορώ να συμφωνήσω να τροποποιούνται με κατοξιοδότηση πράξης. Euh. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των προτάσεων της ακολουθεί μια λογική η οποία μας υποχρεώνει θα έλεγα και μας επιτρέπει ταυτόχρονα να κρατάμε μια κάποια συνεκτικότητα στην πρότασή μας και στην, στον εντοπισμό των κατεξουσιοδότηση πράξεων τις οποίες θα προτείνουμε. Αυτή η λογική μας πρότεινε να φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο κατάλογο και το είπατε εσείς η ίδια, όλα τα άρθρα που επιτρέπουν μία εξαίρεση, 5, 13, 5 λοιπά. Δεν θα τα επαναλάβω όλα, τα αναφερθήκατε σε αυτά εσείς. Όπως επίσης και ορισμένες από τις προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον κανονισμό για τη Μεσόγειο, σχετικά με τις δυνατότητες τις οποίες προβλέπει το άρθρο 26 και 27, και κάποιες προτάσεις επίσης οι οποίες προβλέπουν να τροποποιήσουμε τα παραρτήματα. Υπάρχουν πραγματιορισμένα παραρτήματα τα οποία σήμερα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ γιατί περιμένουμε εμείς το τέλος αυτής της προσπάθειας ευθυγράμμισης η οποία γίνεται και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ξεκινάμε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε εκ των προτέρων να εντοπίσουμε κάποιες από τις προβλέψεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να περάσουμε μετά σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Να πω ότι οι εφαρμοστικές πράξεις προβλέπονται και αυτές, implementing acts, αλλά δεν γίνονται αντικείμενο συγκεκριμένη αναφορά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί θεωρούμε ότι στα πλαίσια αυτών των εφαρμοστικών πράξεων έχουμε να κάνουμε μια αυτόματου τύπου μεταφορά. Εάν όμως ο νομοθέτης απαιτεί ή έστω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο επακριβής στην ποσοστικοποίηση των πράξεων αυτών, <coughs> γιατί όχι θα το κάνουμε. Πάντως επαναλαμβάνω, οι προτάσεις τις οποίες κάνουμε είναι να εντοπίσουμε, να ε, εντοπίσουμε συγγνώμη, τις πράξεις τις οποίες θα εντάξουμε στην κατηγορία των κατεξουσιοδότησιων πράξεων και όλες οι πράξεις τις οποίες δεν αναφέρουμε αυτόματα μετατρέπονται σε εφαρμοστικές. Είμαι στη διάθεσή σας για να μπω στη συζήτηση σε λεπτομέρειες πράξη κατά πράξη. Αλλά παρόλα αυτά ακολουθήσαμε μια λογική η οποία μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τις διαδικασίες οι οποίες ενετάσσονται στην προηγούμενη διαδικασία της επιτροπολογίας και για τις οποίες προτείνουμε να περάσουμε στις κατεξουσιοδότηση πράτης. Η πράξη αυτή είναι η πρώτη η οποία κατετέθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται ε, για το ότι θέλουμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση για την ευθυγράμμιση έτσι ώστε να μην μπλοκάρουμε κάποιες πιθανές αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ληφθούν, να ζητηθούν εν περιπτώσει από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του τίτλου 11 κανονισμού για τη Μεσόγειο. Από τη μία λοιπόν θελήσαμε να σεβαστούμε τον, τις δεσμεύσεις, τις οποίες είχαμε αναλάβει σαν Επιτροπή, δηλαδή την κατάθεση πριν από τον μήνα Νοέμβριο μιας πρότασης για την ευθυγράμμιση. Έχουμε και τον κανονισμό για τη Μεσόγειο που είναι ένας ζών κανονισμό θα έλεγα και που προβλέπει συγκεκριμένες δυνατότητες για τη χορήγηση εξαιρέσεων όταν ακριβώς σέβονται τις διατάξεις και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να μην καθυστερήσουμε και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δεσμεύσουμε εμείς και να απειλήσουμε την ίδια την ύπαρξη όλων αυτών των δυνατοτήτων που προσφέρονται προς τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ροσμπαχ. Ζητώ συγγνώμη που μίλησα έτσι όπως μίλησα στην αρχή, αλλά δεν ήξερα καν ότι είμαι η δεν έχω δει ούτε καν ένα έγγραφο και θα ήμουν ευγνώμων στην ε, γραμματεία αν μπορούσε να μου αποστείλει ό,τι έγγραφα έχει από την Κομισιόν και γενικώ όλα τα όσα αφορούν αυτή την, ε, αυτό το θέμα και θα επανέλθω όσο δυνατόν πιο ε, προετοιμασμένη. Και ζητώ ταπεινά συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Εντάξει. Οπότε Θα μας δώσετε με την ε, γραμματεία ένα χρονοδιάγραμμα και θα το δούμε το θέμα αυτό πάλι στην ε, επόμενη συνεδρία. Ο κύριος Φερέιρα δεν είναι εδώ, δεν θα έρθει. Όχι, δεν θα έρθει ο κύριος Φερέιρα. Ωραία, οπότε θα αναβάλουμε το σημείο του. Άρα πάμε στο επόμενο σημείο και κλεισμένων των θυρών, ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Επιτροπής σχετικά με τις ε, συμφωνίες αλίας. Όποιοι δεν θα συμμετέχουν σε αυτή τη σε παρακαλώ να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Κύριε Ντεπίπερ, παρακαλώ, ελάτε εδώ στο πόντιου.